έχει ζητήσει να μιλήσει ο κύριος Καλινόσκι. Επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένοι από τους τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία ή η βιομηχανία εάν δεν, ε, δεν γίνουν αντικείμενο σωστής διαχείρισης θα αποβούν σε βάρος ε, του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι πόροι αυτοί και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη Βαλτική θάλασσα. Εάν αγνοήσουμε την ανάγκη αυτή, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στους οικονομικούς κλάδους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς και χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Μόνο χάρη μόνο στην βάση διεθνίου συνεργασίας στην έρευνα μαζί με την ρωσική πλευρά είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στι ανάγκες αυτές. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση Τσικλούνα ζήτησε να ζητήσει να μιλήσει ο κύριος Πίτερ Γιάρ. Κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για κάθε νέο μέλος της Ευρωζώνης και έτσι εύχομαι το καλωσόρισες στην, στις καινούργιες χώρες που έχουν ενταχθεί. Επίσης θέλω να επενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν και κριτήρια σταθερότητας τα οποία οφείλουν να τηρούνται. Ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι τα, οι παλαιότερες χώρες μέλη της Ευρωζώνης ε, έχουν την εντύπωση ότι απολαμβάνουν κάποια προνόμια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ισχύει ιδιαίτερα δηλαδή, αυτό για τα κριτήρια σταθερότητας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σύριο Βίρ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη προς το ευρώ και ως εσθονή φυσικά υπερψήφισα την έκθεση για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε και εμείς στη χώρα μας το ευρώ. Εμείς έχουμε μικρό δημόσιο χρέος και έλλειμμα. Είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. υπερψήφισα την έγκριση της έκθεσης και διότι ήθελα να ευχαριστήσω το εσθονικό έθνος. Έχουμε βέβαια προβλήματα με την ανεργία και τους μισθούς και δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Γι' αυτό ελπίζουμε με το ευρώ να τα λύσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αντρική στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ψήφισα υπέρ και θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Εσθονία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να της επιτρέψει να εισέλθει στην Ευρωζώνη από τις αρχές του 2011. Το ευρώ αντιμετωπίζει προκλήσεις σήμερα, αλλά η είσοδός του στην Εσθονία θα πρέπει να μας δείξει ποιες είναι οι προοπτικές που διαθέτει αυτό το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Να πάρουμε σαν υπόδειγμα την εμπειρία της Εσθονίας με όλες τις προσπάθειες που έκανε για να μπει και στην Ένωση και στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα όταν σκεφτούμε ότι η Εσθονία τα κατάφερε όλα αυτά μέσα στην κρίση. Η περίπτωση της Εσθονίας πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες υποψήφιες χώρες μέλη καθώς και τα άλλα μέλη της ε, Ένωσης, ιδίως εκείνα που υποτιμούν τη σημασία που έχουν τα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα σε επεξηγήσει ψήφου στην έκθεση της Αρνέσκη για την απαλλαγή του 2008. Ευχαριστώ. Η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα ήταν πολύ δύσκολη στη συγγραφή της. Παρόμοια για απαλλαγή, για του Συμβουλίου είχε καθυστερήσει μέχρι τον Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επιτηρούμε καλύτερα τις δαπάνες όλων των οργάνων γιατί υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης και είναι δύσκολος ο διάλογος με το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά του δώσαμε απαλλαγή και ελπίζουμε να υπάρξει καλύτερη και περισσότερη συνεργασία μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. Τα έγγραφα που, υποβλήθ, που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πιο ακριβίως προς τις δαπάνες του προϋπολογισμού κάθε οργάνου. Τέλος, η περίφημη Συμφωνία Κυρίων από το 70 πρέπει να αλλάξει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σοβαρές πραγματικό ρόλο στην επιτήρηση των δαπανών του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανησυχώ για τις δηλώσεις που έκανε η Προεδρία του Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν στην Κομισιόν τους προϋπολογισμούς τους πριν από τις Εθνικές Βουλές. Αυτό είναι λάθος και ήταν, δεν ήταν καθόλου σωστό ο κύριος Βαν Ρομπόη να ζητήσει μεταφορά τέτοιων εξουσιών στην Ένωση. Μια τέτοια υποβολή των προϋπολογισμών εκ των προτέρων στην Κομισιόν θα αποτελούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και ελπίζω να αγνοηθούν όλες αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Βαν Ρόμποϊ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Πρώτα οι εθνικές βουλές θα εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς. Για ορισμένες χώρες που έχουν προβλήματα, δεν λέω, αλλά όχι για χώρες σαν το ΙΤΑΒ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λάτφορντ έχει ζητήσει να μιλήσει για επεξήγηση ψήφου. Κύριο Σινκλέρ. Uh, Κυρία um, Ευχαριστώ. Εγώ κατεψήφισα την έκθεση αυτή. Όχι επειδή δεν πιστεύω στο θέμα της, δηλαδή στις ποινικέ ε, διαδικασίες και στην απαραίτητη ε, ε, προσέγγιση τους, αλλά αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι η συμπερίληψη της ECHR που ήδη έχει συνυπογράψει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί την οδό αυτή που ακολουθεί. Ε, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι αυτό. Είναι άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση του να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος. Οι εθνικές κυβερνήσεις όμως αντιτάσσονται και είπαμε ότι δεν πρόκειται να, γίνει ευρωπαϊκό, ε, να υπάρξει ευρωπαϊκό κράτος. Εγώ και οι συνάδελφοί μου του Βρετανικού Ανεξάρτητου Κόμματος απέσχομαι, όχι, ότι δεν, όχι επειδή δεν χρειάζεται να υπάρχουν μεταφράσεις των διαφόρων ποινικών διαδικασιών για όσου άγονται ενώπιον αλλοδαπών δικαστηριών, αλλά δεν θέλουμε να μπει στο πρόγραμμα τη Στοκόλμη και την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων. Όπως είπαμε και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, αυτά σημαίνουν ανατροπή των ε, από αιώνων ισχυόντων κανόνων για την προστασία του ατόμου σε περίπτωση σύλληψη και ανάκριση κτλ. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για εντολέ κατασχέσεων κλπ. Όσοι πιστεύουν ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να έχουν τα δικαιώματα να προστατεύουν του πολίτε του θα πρέπει να είναι αντίθετο με την εναρμόνιση των νομικών συστημάτων και του πρόγραμμα Στοχόλμη. Ωραία. Έχουμε τώρα την έκθεση Μπάουερ η οποία απορρίφθηκε. Οι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν παρόλα αυτά. Αν θέλετε το λόγο, έχουμε την κυρία Αντρικίνε και την κυρία Σενκλέρ. Παρακαλώ. Κυρία Αντρικίνε. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την έκθεση Σούριαν για θέματα δημοσιονομικά. ο πρόεδρος. Κύριε Ανδρικίνε, μιλάμε για την έκθεση Bauer, η οποία απορρίφθηκε. Αν θέλετε να παρέμβετε για την έκθεση Σούριαν, μπορείτε να παρέμβετε γραπτός, διότι πρόκειται για μία ε, έκθεση η οποία θα περάσει με απλουστευμένη διαδικασία, επομένως μπορείτε να μας δώσετε τη δήλωσή σας γραπτός. Έχουμε όμως την έκθεση Bauer, η οποία απορρίφθηκε. Η κυρία Σινκλέρ, παρακαλώ. Thank uh, um, Ευχαριστώ. Και εγώ ψηφίσα για την απόρριψη της έκθεσης αυτής. Εκπροσωπώ τα West Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις χειρότερες περιφέρειες ως προς την ανεργία. Όπως και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι προσπαθούν να ανοίξουν μια επιχείρηση, μικρομεσαία ή μικρή επιχείρηση, και εδώ πρόκειται για επίθεση κατά αυτών των προσπαθειών. Η κατάσταση των μικρομεσαίων και ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων δεν είναι καθόλου ευχάριστη ως προς την νομοθεσία που ισχύει. Υπάρχει υπερβολική νομοθεσία. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να μην εφαρμόζονται συνεχώς και καινούργιοι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις γιατί αυτό αυξάνει το βάρος της διοίκησής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σουλάμι, όχι. Ντόρφμαν, παρόν, όχι, απορρίπτεται. Ο κύριος Μαστέλα είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω ότι είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων καταναλωτών να γνωρίζουν τι περιλαμβάνεται στα ε, ε προϊόντα που καταναλώνουν. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει περισσότερο για τα θέματα αυτά. Βέβαια, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει νομική ασφάλεια για όσους συμμετέχουν στην ε, διατροφική αλυσίδα και στην, ε, στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων και να υπάρχει ασφάλεια για την υγεία των καταναλωτών στα διατροφικά προϊόντα. Απ' τη μια έχουμε τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία και να έχουμε νομοθετική απλούστευση. Κατ' εμέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεραπλούστευσε τα πράγματα. Υποστηρίζω την πρόταση τη ηγήτρια για τα διατροφικά προφίλ, τα οποία ε, διευκρινίζονται μεν με πολύ ενδολοχή τρόπο, αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικέ γνωμοδοτήσει που να τα εγκρίνουν. Με εκπλήσει το γεγονός ότι εκπονήθηκε μια τέτοια έκθεση χωρίς να ανατρέξουμε στους εμπειρογνώμονε ε, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να ε, ξεκινάει ένα διατροφικό προφίλ. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί τα επιστημονικά στοιχεία και θα ξεκινάει η έρευνα σε κάθε κράτος μέλος. Και τώρα είστε εγγεγραμμένοι, θα μιλήσετε, μην ανησυχείτε, ο Πίτερ Ζάρ. Βεβαίω οι καταναλωτέ, κύριε Πρόεδρε, έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι περιλαμβάνεται στα τρόφιμα. Όποιο πιστεύει όμω ότι με τη νέα αυτή νομοθεσία θα οδηγήσει σε υγιέστερη διατροφή των καταναλωτών, κάνει λάθο. Αυτό που χρειάζεται είναι σωστή ενημέρωση, εκπαίδευση και για τους ενηλίκου και για τα παιδιά. Όποιο ε, διατρέφεται από πολλές πηγές, όποιος ασκείται τακτικά και δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τις σοκολάτες αν αυτές του αρέσουν για παράδειγμα. Μπρεζίνα. Απόν. Ο κύριος Μάριο Πυρίλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την έκθεση Σόμορ καταψήφισα τις τροπολογίες που εισαγάγουν το ε, λεγόμενο σύστημα του σηματοδότη. Θεωρώ ότι το να αναφέρονται τα λίπη, τα άλατα, τα σάκχαρα, τα κορεσμένα λίπη και η ενεργειακή απόδοση ε, μέσω ενός απλού συστήματος ε, με χρώματα δεν δίνει στον καταναλωτή τις σωστές πληροφορίες. Ελοχεύει ο πραγματικός κίνδυνος να να τιμωρήσουμε έτοιμα γεύματα, όπως για παράδειγμα την κατεψυγμένη πίτσα, η οποία θα έχει μια κόκκινη ετικέτα στην συσκευασία γιατί περιλαμβάνει τυρί. Ο σηματοδότης ε, παραδόξως ευνοεί προϊόντα τα οποία δεν είναι και τόσο υγιεινά σε σχέση με πιο ποιοτικά προβλήματα, προϊόντα. Δεν είμαι υπέρ λοιπόν της ένδειξης επίσης ε, στις ε, ετικέτες της ε, θερμιδικής περιεκτικότητας σε είναι ποτέ, συμπεριλαμβανομένου και του ίνου και θεωρώ ότι δεν λάβαμε παρκώς υπόψη στα θέματα της προέλευσης των τροφίμων. Ευχαριστούμε τον κύριο Πυρίλο. Κυρία Όβιρ Σύρη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 Και για την έκθεση της Κιασόμερ Σόμερ θέλω να πω ότι αναγνωρίζω το έργο που επετέλεσε και προτιμώ να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι κανόνες και έτσι για τον λόγο αυτό υποστηρίζω την έκθεση. Την επιστήριξα δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επισημαίνεται ο αριθμός των θερμίδων για παράδειγμα σε κάποιο ποτό αλλά δεν συμφωνώ με το σύστημα του σηματοδότη που νομίζω ότι είναι εν τέλει πολύ υποκειμενικό είναι υποκειμενικό και ταυτόχρονα δεν προσφέρει επαρκείς πληροφορίες για μια σωστή εξισορρόπηση διατροφής όταν μιλούμε για χρώματα κόκκινα, κίτρινα, πράσινα δίνουμε απλώς μια πληροφορία σχετικά με το πώς ε, αντιλαμβάνονται την αξία των τροφίμων αυτών οι καταναλωτές. Εδώ έχουμε επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Σόμερ. Έχω και για την έκθεση της κυρίας Πάουερ να πω κάτι. Εγώ σήκωσα το χέρι μου εγκαίρος εμείς δεν λάβαμε σχετικό έτοιμο. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο τώρα για την έκθεση Bauer, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έκανε σημαντικό έργο η κυρία Μπάουερ και εγώ ήμουν μέλος της ε, Επιτροπής και είδα τι δουλειά έκανε. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα να περιληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι γιατί αυτοί καλύπτονται από τον κανονισμό 51. Έτσι λοιπόν εγώ δεν υποστήριξα την απόσυρση της έκθεσης. Καρινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η βασική ιδέα του ψηφίσματος αυτού είναι να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπως ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει η ίδια σήμανση των τροφίμων για να είναι τα πράγματα πιο σαφή για τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες. Χάρη σε αυτή την εναρμονισμένη λύση και εναρμονισμένους κανόνες για την ετικετοποίηση των τροφίμων θα μπορούν πιο εύκολα οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες να γνωρίζουν τι καταναλώνουν και τι ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να υπάρχουν ή αλλεργιογόνα για να μην τα καταναλώνουν κατά λάθο. Έτσι θα απλοποιηθεί η λειτουργία της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή βέβαια στη σήμανση των τροφίμων χωρίς να υπάρξει μεταβατική περίοδος θα κατέληγε σε σημαντικούς κινδύνους για τους παραγωγούς. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο που εγκρίναμε σήμερα. Πρέπει να πληροφορούμε σωστά τους καταναλωτάς και τα καταναλωτρίας. Και να είναι η πληροφόρηση αυτή εύληπτη Πρέπει όμως να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ της σημαντικής και της ασήμαντης πληροφόρησης για να προασπίσουμε έτσι τα συμφέροντα των καταναλωτών και να δημιουργήσουμε έτσι ένα σύστημα που ενθαρρύνει τη χορήγηση πρόσθετων πληροφοριών. Είναι κάτι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την καλή υγεία όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Ο κανονισμός προβλέπει καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη φιλοπληροφόρηση των καταναλωτών ώστε να αποφεύγεται η παχυσαρκία. Και ταυτόχρονα μια απογραφειοκρατικοποίηση. Με την απόφαση που λάβαμε σήμερα θα έχουμε πράγματι πολλές πληροφορίες διαθέσιμες για τον καταναλωτή. Τώρα αν θα είναι αποτελεσματικό αυτό θα φανεί με το μέλλον. Αλλά θέλω να επισημάνω οπωσδήποτε ότι η αλυσίδα καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη, καλύτερη επισήμαση, καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη υγεία δεν είναι δεδομένη. Θα χρειαστεί λοιπόν το Κοινοβούλιο να κάνει ακόμα μεγάλη προσπάθεια πληροφόρησης και κυρίως τα σχολεία. Σε ό,τι αφορά την απογραφειοκρατικοποίηση, εδώ πετύχαμε ακριβώ το αντίθετο. Εάν σκεφτώ ότι για παράδειγμα εξακολουθούμε να έχουμε τα λεγόμενα διατροφικά προφίλ, ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με την προέλευση, φορτώνουμε λοιπόν και άλλη γραφειοκρατία στον πολίτη και νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν θα την παίρνει καν υπόψη του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ και άλλοι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την έκθεση Σόμερ στο τελική ψηφοφορία γιατί θεωρούμε ότι επετεύχθη κάποια πρόοδος σε δύο θέματα, στη χώρα προέλευσης και στην επισήμανση στη συσκευασία. Έχουμε βέβαια παράλληλα αυτά πολλές επιφυλάξεις για την ε, υπερψήφιση της ε, κατάργησης εθνικών εθελοντικών ε, προγραμμάτων επισήμασης όπως το πρόγραμμα που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για εθελοντικά προγράμματα και κατά πώς φαίνεται αρέσουν στους καταναλωτές. Θα δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο για την διατήρηση αυτών των εθνικών προγραμμάτων, αλλά ελπίζουμε ότι αν φτάσουμε σε δεύτερη ανάγνωση, αν δεν μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία ανά την Ευρώπη για τους σηματοδότες, τουλάχιστον τα κράτη-μέλη που έχουν εθνικά προγράμματα τα οποία λειτουργούν σωστά και είναι κατανοητά από τους πολίτες, θα, να πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ την κυρία Μακάουα, Μακά... Ο κύριος Μπάτεν για την οικονομική διακυβέρνηση τώρα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταψήφισα το ψήφισμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική συνέπεια, αντικατοπτρίζει τον τρόπο ε, και την οδό προς την οποία κατευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά. Όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί, ο κύριος Μπαρόσο και ε, οι επικεφαλείς των περισσότερων ε, πολιτικών ομάδων μας είπαν ότι αυτό ακριβώς θέλουν. Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ως μία κρίση που ε, μας βοηθά να επεκτείνουμε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ εκπροσωπώ το City του Λονδίνου που κινδυνεύει να καταστραφεί από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανική οικονομία θα καταστραφεί στο σύνολό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λογικό λοιπόν στοιχείο που περιελάμβανε ήταν η έκθεση του κυρίου Πάιπερ που επιτρέπει στη κράτη-μέλη να ε, φύγουν από το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Νόμισμα. Εγώ την υπερψήφισα αυτή την τροπολογία, αλλά δυστυχώς απορρίφθηκε. Θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ τους πάντες.